Τα πρακτικά θα τα βρείτε λοιπόν δημοσιευμένα και σύμφωνα θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου την Τρίτη θα υπογράψουμε έξι πράξει που εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78. Δημοσιεύονται επίση. Να περάσουμε στο, σχέδιο, στο